Εκτά. Περνάμε τώρα στη σειρά των εργασιών μας. Καταρχάς, η τελική ημερήσια διάταξη, όπως καθορίστηκε την Πέμπτη από την διάσκεψη των Προέδρων, σύμφωνα με το άρθρο 149, έχει ήδη διανεμηθεί. Δεν έχω λάβει κάποιες αιτήσει τροποποίησης της ημερήσιας διάταξης. Έτσι λοιπόν παραμένει ως έχει. Σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει η πανηγυρική συνεδρίαση. Συνάδελφοι, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια, ένα κενό έδρανο εδώ. Ανήκει σε ένα από τα πολιτικά κόμματα της Γαλλίας, την κυρία Μαρίν Λεπέν. Είναι απούσα η κυρία Μαρίν Λεπέν, όχι επειδή υπάρχουν προβλήματα στα βελγικά αεροδρόμια, αλλά γιατί έχει ταξιδέψει στη Μόσχα. Σύμφωνα με τον τύπο πηγαίνει στη Μόσχα για να πάρει πιστώσεις από τους συμμάχους της, τους Ρώσους. Αλλά δεν είναι μόνο χρηματικό το θέμα. Πηγαίνει εκεί γιατί δέχεται οδηγίες και θα ακούσουμε τις οδηγίες αυτές αργότερα ε, και γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσω από τις γαλλικές αρχές ε, να εξετάσουν προσεκτικά τέτοιου είδους περίεργες και ύποπτες πολιτικές συμπεριφορές. Ε, δεν μου φάνηκε το θέμα αυτό ιδιαίτερα στην ημερήσια διάταξη, λέει ο Πρόεδρος. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή του συναδέλφου ότι η Μαρίν Λεπέν είναι στο Παρίσι, ότι αν ο συνάδελφος θέλει να ενημερωθεί για τις σχέσεις τις οποίες έχουμε με τον πρόεδρο της Ρωσικής Δούμα, με τον οποίο συζητάμε σε ετήσια βάση, τον πρόεδρο Ναρίσκιν. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με ιστορίες για χρηματοδοτήσεις, αλλά έχει σχέση με την πολιτική και τις σχέσεις που έχουμε σε σταθερή βάση με τους Ρώσους συναδέλφους εδώ και 20 χρόνια. Λοιπόν, σας παρακαλώ αγαπητέ συνάδελφε, ε, σταματήστε να λέτε ότι σας περνάει από το νου και να ψαρεύετε πληροφορίες σε θολά νερά και παρακαλώ να παραμείνετε ένας τίμιος βουλευτής και πέραν αυτού τίποτα. Κοιτάξτε συνάδελφοι, το θέμα δεν είναι στην ημερήσια διάταξη. Έχει δει στο λόγο άλλος ένας συνάδελφος. Αγαπητοί συνάδελφοι, και εγώ θα ήθελα να ζητήσω από τη διάσκεψη των Προέδρων να εξετάσει τη δυνατότητα να θεωρήσει πρόβλημα σύγκρουσης συμφερόντων για οποιοδήποτε πολιτικό ο οποίος παίρνει δάνεια από το εξωτερικό. Αυτό ισχύει για το κόμμα, το εθνικό μέτωπο στη Γαλλία. Ζητώ από το Προεδρείο να εξετάσει το θέμα αυτό πάρα πολύ σοβαρά. Κύριε Μποστινάρο, το θέμα αυτό δεν είναι στην ημερήσια διάταξη. Αν θέλει ο πρόεδρος της πολιτικής σας ομάδας μπορεί να το θέσει στην επόμενη συνεδρίαση της διάσκεψης των πρόεδρων. Λοιπόν, τελειώνει εδώ το θέμα. Ξεκινάει η επίσημη συνεδρίαση, η πανηγυρική συνεδρίαση. Το θέμα, όπως είπα, δεν είναι στην ημερήσια διάταξη. Έθεσε το θέμα ένας βουλευτής, απάντησε ένας άλλος βουλευτής. Τώρα θα πρέπει να επιτρέψουμε την εκκίνηση της πανηγυρικής συνεδρίασης και να ακούσουμε προσεκτικά τον φιλοξενούμενό μας, τον κύριο Μπαν Κιμούν. Διακόπτουμε για ένα λεπτό για να δώσουμε τη δυνατότητα στον πρόεδρο Σούλτς και στον πρόεδρο Κίμουν να μπουν στην αίθουσα.

Αξιότιμη Γενική Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, είναι μεγάλη μας χαρά να σας καλωσορίσουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκ νέου. Αξιότιμη κυρία Μπαν, και προς εσάς ε, σας, ε, κυρία Μπαν, σας καλωσορίζουμε και εσάς εδώ που συνοδεύσατε